Um, ladies and gentlemen, I know Έρχονται και άλλοι συνάδελφοι σιγά σιγά κυρίες και κύριοι. Χριστούγεννα έρχονται. Να καλωσορίσω ωστόσο τους, ε, τον κύριο Μπερνατόνης και τον κύριο Μπαρακάουσκας από την Προεδρία και θα τους ζητήσω να μας δώσουν μια εικόνα των δραστηριοτήτων της ε, Προεδρίας. Φαντάζομαι ότι θα πούν και το είδαμε. Ήταν μια θετική Προεδρία. Κάποια πράγματα δεν έκλεισαν δεν ξέρω τώρα, προστασία δεδομένων, φοβάμαι να το πω. Όποτε το βλέπω όπου το θίγω δημιουργούνται ζητήματα αλλά και σε άλλα, σε άλλα ζητήματα την κατάσχεση προϊόντων εγκρήματος και άλλη υπήρξε μεγάλη πρόοδος είμαι σίγουρος πάντως ότι θα υπάρξουν σχόλια Κύριε Υπουργέ Κύριε Υπουργέ Μπερνατώνης έχετε το λόγο Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την ευκαιρία να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της προεδρίας μας στον τομέα της δικαιοσύνη. Παρότι αυτό ήταν η πρώτη προεδρία της Λιθουανίας στο Συμβούλιο, το έργο ήταν πολύ θετικό και όλα τα μέλη της Προεδρίας ήθελαν να δείξουν ότι θα πετύχαιναν αυτά που είχαν παρουσιάσει ε, τον Ιούλιο και βεβαίως πολλά από αυτά που είπαμε δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη βοήθεια των άλλων οργάνων της Ένωσης. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και εσάς ε, κυρίως για την συνεργασία και βοήθεια που δείξατε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε, ε, να προχωρήσουμε ταχύτερα ακόμα περισσότερο. Ελπίζουμε ότι δεν σας ε, απογοήτευσαν τα αποτελέσματα της Προεδρίας και θέλω να τα παρουσιάσω εντάχει. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας η έμφαση δόθηκε σε τρεις τομείς. Να δημιουργηθεί μια ανοιχτή αξιόπιστη Ευρώπη και στον τομέα της δικαιοσύνη υιοθετήσαμε μέτρα που θα προκαθιστούσαν την εμπιστοσύνη στην Ένωση. Θα εξασφάλιζαν την δημοσιονομική σταθερότητα, θα ενίσχυαν την οικονομική και νομισματική ένωση και θα παρουσίαζαν ασφάλεια, τα, θα προσθέτουμε ασφάλεια τα συμφέροντα της Ένωσης. Επίσης, Τρία συμπεράσματα δόθηκαν στην ενίσχυση των σχέσεων της Ένωσης με, τις τέσσερις, ε, με, με τους ε, τρίτους εταίρους μας, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης Ευρώπης με αποτελεσματική οικονομία και διαχείριση της οικονομίας της. Δουλέψαμε για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον τομέα της ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η πρόοδος στον τομέα της δικαιοσύνης ε, δημιούργησε μια αξιόπιστη Ευρώπη. Το θέμα ήταν η παγίωση της ασφάλειας των δημοσιονομικών συμφέροντων της Ένωσης με μέτρα ποινικού δικαίου. Εδώ είχαμε και την βελτίωση φυστάμενων πρωτοβουλειών και τη δημιουργία νέων. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε μια αξιόπιστη Ευρώπη, κυρίως με την οδηγία για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη. Θέλουμε τα εργαλεία να είναι σημαντικά για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του ευρώ και άλλων οργάνων και, άλλο, άλλων νομισμάτων από την, από, την παραχάραξη. Με χαρά μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τις ε, διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο με μια κοινή θέση. Οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο στην πρώτη αυτή πιστεύουμε ότι θα είναι επικοδομητικές και ε, επιτυχής και ότι θα υπάρξει συμφωνία ε, σε πρώτη ανάγνωση. Ένα άλλο σημείο προτεραιότητας είναι η οδηγία για την κατάσχεση προϊόντων ποινικών ποινικών αδικημα... Ε, αδικημάτων. Στην Προεδρία μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο στην πρόταση αυτή και νομίζω η έγκρισή της είναι ένα τεράστιο βήμα για να εξασφαλίσουμε ότι το έγκλημα δεν θα αποδίδει. Παρότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες λόγω των διαφορών μεταξύ των θέσεων των θεσμικών οργάνων, είμαστε ικανοποιημένοι ότι μπορέσαμε να πετύχουμε κοινή συμφωνία για το κείμενο της νομικής ε, του νομικού κειμένου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια της Επιτροπής σας κύριε Μακοβέ για την ε, επινόηση ε, καλών λύσεων και θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση διότι μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επετεύχθηκε συμφωνία για, την ευρωπαϊκή, για το ευρωπαϊκό ένταλμα που επιτρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, ε, ε, ένταλμα έρευνας μεταξύ, που επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ των ε, υποχρεώσεων προστασίας και των υποχρεώσεων ασφάλειας. Κάτι που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση με επιτυχία των ποινικών ανακρίσεων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια από την Επιτροπή σας για την αναζήτηση συμφωνίας στο κείμενο αυτό. Ελπίζουμε ότι η οδηγία θα υιοθετηθεί στο εγγύς μέλλον. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας ε, ξεκινήσαμε επίσης τριμερείς διαλόγους για την πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και Συμβουλίου για τις ποινικέ κυρώσεις για το, την ε, ε, ε, χειραγώγηση αγοράς και το inside dealing. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας έγιναν εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι προσπάθειες, ε, συνεχίστηκαν οι εργασίες στο Συμβούλιο για το νομοθετικό κείμενο και θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το, την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας στις διαπραγματεύσεις και να ευχαριστήσω τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την ε, αναζήτηση λύσεων. Ελπίζω ότι στο τέλος της προεδρίας θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία για τα βασικά εργαλεία του σχεδίου νομοθετικού κειμένου Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας επίσης δώσαμε μεγάλη σημασία στις προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ποινικής Δικαιοσύνης και την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Οι προτάσει που συζητήθηκαν τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη έδειξε ότι η πλειοψηφία των Υπουργών υποστήριξαν την ιδέα της Ευρωπαϊκής της Αγγελικής Αρχής, ωστόσο θεώρησαν ότι η πρόταση πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Σε ένα σύντοστο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρουσίαση της πρότασης νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει σε πολλά από τα θέματα που συζητήθηκαν ε, όπως δομή, αρμοδιότητες. Παρότι είναι νωρίς να πούμε ότι το θα ολοκληρωθεί σύντομα το, το, σύστημα. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του γραφείου της αγγελίας σταδιακά θα, θα υλοποιηθούν. Το Σεπτέμβριο του 2013 με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου οργανώσαμε, σας το θυμίζω αυτό, μια επιτυχή συνάντηση για την ε, εξέταση της πρότασης στο μέλλον. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό υπογραμμίστηκε και από την πλειοψηφία των Υπουργών Δικαιοσύνης. Η Επιτροπή νομίζω υποστηρίζει τη θέση που εκφράστηκε στην ανακοίνωση της 27ης Νοεμβρίου, κάτι θετικό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργείται βάσει του Eurojust με την πρόταση ε, της, συνεργασίας στα ποινικά ζητήματα. Με δεδομένη την αύξηση του διασυνοριακού εγκλήματος είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του Eurojust. Οι συζητήσει τη ομάδα εργασία για το θέμα αυτό ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο με την ανάλυση των τριών πρώτων κεφαλαίων του κανονισμού. Η δουλειά, πιστεύουμε, θα βοηθήσει στην ε, περαιτέρω ολοκλήρωση των συζητήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμη δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ε, προσοχή στην προστασία των πολιτών και ότι το 2013 ήταν ε, το έτος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαίου πολίτη, πολίτη, η Προεδρία ασχολήθηκε για τα θέματα ισότητας ευκαιριών, διάκρισης, στο πλαίσιο αυτό θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου με την τελική συμφωνία που επιτεύχθηκε για, το νέα, για τα νέα χρηματοοικονομικά προγράμματα και την υλοποίηση των στόχων αυτών. Το πρόγραμμα Justice και το πρόγραμμα Ισότητας και Ιθαγένειας. Μας ικανοποιεί το ότι το Συμβούλιο συμφώνησε με το Κοινοβούλιο στις δύο αυτές προτάσεις. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις που εξασφάλισαν ότι η πρόταση μπορεί να εγκριθεί πριν το τέλος ε, του έτους. Επίσης μας ικανοποίησε ότι εγκρίθηκαν οι προτάσεις στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου και χτες, 16 Δεκεμβρίου, επίσημα και από το Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κίνγκα Γκούντς του εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την επικοδομητική συνεργασία στην επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών. Η ανάμνηση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το έτος Ευρωπαίου Πολίτη 2013 εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο χτες και το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών της Ευρώπης για τα δικαιώματά τους και για τη δυνατότητα να το εφαρμόζουν σε καθημερινή ε, βάση χωρίς ε, εμπόδια. Τα συμπεράσματα αυτά ε, δίνουν έμφαση στους στόχους μείωσης των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκουμένων και φοιτητών για την προστασία των ευάλωτων ομάδων πολιτών της Ένωσης για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας της πληροφορίας και την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία. Ταυτόχρονα η μείωση, με μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, η έμφαση στο πολίτη επέτρεψε να οργανώσουμε στο Βίνιους μια διάσκεψη για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη στις 12 Δεκεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου έγινε μια διάσκεψη στο Κοινοβούλιο της Λιθουανίας. Το γεγονός, ε, το γεγονός αυτό ήταν μια ευκαιρία να δούμε ό,τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια του έτους για την βελτίωση των, της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και για να παράσχει στην Ένωση για να παράσχει περαιτέρω καθηγητή γραμμή. Με, με πρωτοβουλία της Λιθουανικής Προεδρίας κλήθηκαν και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών ε, φορέων. Μια ευκαιρία να δουν πώς είναι η κατάσταση πραγματικά, να δούμε πώς είναι η κατάσταση πραγματικά για τους πολίτες της Ένωσης και να δούμε τις προοπτικές της ηθαγένεια της Ένωσης από αυτό το πρίσμα. Συνεχίζουμε το έργο για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της Προεδρία μας η Επιτροπή υπέβαλε ερώτημα στο Δικαστήριο της Ένωσης ζητώντας την άποψή του για το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Κάτω από την παρότριση της πλειοψηφίας των κρατών μελών, η Προεδρία έστειλε επιστολή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κυρία Ρέντινγκ, ζητώντας από την Επιτροπή να μας δώσει ε, ενοποιημένη εκδοχή των εσωτερικ, του εσωτερικού κανονισμού. Απάντησε ωστόσο ο, η Επιτροπή ότι αυτό το κάνει μετά τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Παρά τα το Συμβούλιο συνέχισε να δουλεύει σε διάφορες διαστάσεις του κανονισμού. Στις 2 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο εξέδωσε δύο ομάδες συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα συμπεράσματα της πρώτης ομάδας είχαν στόχο την αξιολόγηση, την αξιολόγηση της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Η Προεδρία με, είχε στόχο να συμβάλλει στην περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών, παρουσιάζοντας προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού δημιουργίας της ΦΡΑ, της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Συνολικά κρίθηκε θετική η δουλειά της υπηρεσίας αυτής, ενώ ετοιμάστηκαν και συμπεράσματα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υπηρεσία και της καλύτερης επικοινωνίας τους ε, με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που ετοίμασε η Προεδρία και, συμφω... και επί των οποίων συμφώνησαν το Δεκέμβριο είχαν στόχο την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα αυτά έχουν ως στόχο να αυξήσουν την επίγνωση για τα εγκλήματα μίσους που ενθάρρει και παροτρύνοντας την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτάσεων για την καταπολέμηση τέτοιων μορφών βίας στα κράτη-μέλη και πανενωσιακά. Η διάσκεψη στην οποία η Προεδρία με την ΦΡΑ ε, οργάνωσαν στις 12 και 13 Νοεμβρίου έθεσε τα θεμέλια των συμπερασμάτων αυτών του Συμβουλίου. Το προήμιο των συμπερασμάτων περιλαμβάνει μνήμα στην ιστορική μνήμη της Ευρώπης και καταδίκη όλων, όλων των εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της και εγκλημάτων πολέμου, που ε, μεταξύ άλλων και από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Προχωρώ δημιουργία μιας μεγαλύτερης Ευρώπης. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα νομοθετικά κείμενα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Το πακέτο μεταρρύθμισης των, της, της προστασίας δεδομένων είναι μια σύνθετη διαδικασία με στόχο την εξισορρόπηση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη. Το πακέτο μεταρρύθμισης ε, των ε, προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα της ε, Προεδρίας. Συνεργαστήκαμε με τους Ιρλανδούς και με τους εμπειρογνώμονες σε όλα τα επίπεδα. Το πακέτο μεταρρύθμισης προστασίας των δεδομένων αναλύθηκε για 20 ημέρες τουλάχιστον και συμπεριελήφθη και στις άτυπες συναντήσεις τον Ιούλιο στο Βίλνιους και στα Συμβούλια Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανακύψει ένας ενιαίος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και να προβάλλουμε μία μονοθυριδική προσέγγιση. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό και θα ήθελα να τονίσω ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση Υπουργών του Οκτωβρίου, να φτάσουμε σε συνένεση ως προς το μονοθυριδικό πρότυπο, το οποίο είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που ακόμα δεν έχει επιληθεί σε υπουργικό επίπεδο. Ε, προωθήθηκε εντατική εργασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, όμως οι Υπουργοί δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ως προς το μηχανισμό. Ανέκυψαν νομικής υφής ζητήματα, ιδιαίτερα ως προς τη μονοθυριδική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο θα επιδίνωνε την κατάσταση των πολιτών και θα υπέσκαπτε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό οι Υπουργοί ε, δεν θέλησαν να λάβουν απόφαση με τέτοια σπουδή. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε έναν κανονισμό υψηλής ποιότητας που θα, και που θα αποτελέσει πραγματικά προστιθέμενη αξία για την εσωτερική αγορά και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Η ελληνική προεδρία θα προωθήσει το θέμα και ελπίζω να επέλθει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη μπορεί να αρχίσει ε, συζητήσεις με το Συμβούλιο. Τέλος, Θέλησαμε να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή Ευρώπη, δηλαδή παρά τις τρέχουσες προκλήσεις η Ευρώπη παραμένει ανοιχτή. Το τελευταίο εξάμεινο προωθήσαμε τη συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσα στα πλαίσια λοιπόν ε, των ομολόγων μας και στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών τον Οκτώβριο προωθήσαμε αυτό το θέμα. Εγκρίναμε μια κοινή δήλωση με συγκεκριμένα βήματα για στενότερη συνεργασία σε επίπεδο δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρων. Αυτή η πρώτη προσέγγιση ήταν πολύ ευεργετική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ε, χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προωθηθεί περαιτέρω αυτή η συνεργασία τον Ιούλιο υπέβαλα τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε ότι ίσως θα πρέπει να εργαστούμε και σε θέματα και για θέματα που δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ατζέντα μας. Ε, εδώ αναφέρομαι στη δράση της NSA και στη συλλογή πληροφοριών μέσα στα πλαίσια των υποκλοπών. Εδώ ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα και αυτό αφορά θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που παραβιάζονται, δηλαδή παραβίαση του ιδιωτικού βίου των Ευρωπαίων πολιτών μέσα στα πλαίσια της ε, ηλεκτρονικής κατασκοπίας. Προωθήσαμε το διάλογο με τις ΗΠΑ για να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ για την προστασία δεδομένων. Θα, θέλουν, θα θέλαμε να λάβουμε θετικά μηνύματα από τη ΣΥΠΑ, γιατί πρόκειται για άνηση μεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών και Αμερικανών. Μετά από αιτήματα προώθησης πληροφοριών, μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης ε, της πολιτικής ε, πληροφοριών των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να συνεισφέρουν μέσα στα πλαίσια του Αμερικανικού Προγράμματος Εποπτείας που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο. Υποβάλαμε τα αιτήματά μας στις ΙΠΑ από το Δεκέμβριο και μετά και θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Η Προεδρία έλαβε υπόψη και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μέσα στα πλαίσια των βασικών ελευθεριών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων που θα λήξει σύντομα. Μέσα στα πλαίσια της συνάντησης του Βίλνιου στον Ιούλιο ξεκινήσαμε ένα πολιτικό διάλογο επί του θέματος και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους για κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων γραπτός. Κατά τη Λιθουανική Προεδρία προωθήσαμε συζητήσει σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αποφανθήκαμε το Δεκέμβριο. Επίσης προτιμάσαμε τις ε, προκαταρκτικές προτάσεις των κρατών μελών και η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει περαιτέρω το θέμα. Πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ορίσουν τις ε, μελλοντικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές μέσα στα πλαίσια των βασικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις πρωτοβουλίες για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Το Συμβούλιο ε, δέχτηκε τις βασικές προτεραιότητες και θα προωθήσουμε και τον κανονισμό για τις διαδικασίες περί αφαιρεγγιότητας. Ορίσαμε κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω συζητήσεις. Το Δεκέμβριο επίσης εγκρίναμε μία κοινή θέση για τροποποίηση του κανονισμού των Βρυξελών 1 και προωθήσαμε συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Μέσο Πολίσεων. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτά είναι τα βασικά ε, συμπεράσματα στον τομέα της δικαιοσύνης. Πέραν όμως από τις πρωτοβουλίες επεξεργαζόμαστε και άλλα ζητήματα για να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Το τελευταίο εξάμεινο ε, αποτελεί ένα νέο ορόσημο το οποίο ορίζει τις, ε, τις συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα στα πλαίσια από πλευράς Προεδρίας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία και βοήθειά σας τους τελευταίους μήνες. Ελπίζω μέχρι το τέλος της Προεδρίας να προωθήσουμε κοινούς κανόνες και θα προωθήσουμε τη συνεργασία μας με βάση θέματα που θα προωθήσει η Ελληνική Προεδρία. Είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις σε ερωτήσεις. Σίγουρα ήταν μια περιεκτικότατη παρουσίαση της Λιθουανικής Προεδρίας, όμως δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η παρουσίαση, διότι θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Μπαρακάουσκα να μας κάνει την δική του παρουσίαση για το δικό του απολογισμό. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που με καλέσατε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συνεχίσω την παρουσίαση του συναδέλφου μου, Υπουργού Δικαιοσύνη τη Λιθουανίας, κ. Μπερνατώνης και να σας παρουσιάσω τη δουλειά που κάναμε στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Πρωτού αρχίσω, ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα την Επιτροπή αυτή, καθώς και όλους τους εισηγητές της για τον επικοδομητικό διάλογο και την καρποφορό συνεργασία. Ήταν πραγματικά επιτυχημένη η συνεργασία μας. Θα ήθελα να αρχίσω με τα οριζόντια ζητήματα και συγκεκριμένα με το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2004 έως το 2020. Εργαστήκαμε πάνω σε τέσσερις κανονισμούς στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Ε, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις και τριμερείς διάλογοι τους τελευταίους έξι μήνες εντατικότατα. Και η δουλειά συνεχίζεται. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία και ε, για δημοσιονομικά θέματα στον τομέα των, ε, της εσωτερικής ασφάλειας και για τους ε, εναπομείνοντας δύο κανονισμούς. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω η τελευταία συμφωνία για τα έγγραφα αυτά επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα. Η συμφωνία λοιπόν επετεύχθη και να είστε σίγουροι δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση και κανένα εμπόδιο στη χρηματοδότηση των εσωτερικών υποθέσεων από το 2014. Όπως ανέφερε ο συναδελφός μου, μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, προωθήσαμε τις ε, συζητήσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της δικαιοσύνης και των πολιτικών υποθέσεων. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα επιτύχαμε. Θα ήθελα να πω όμως ότι όλα τα κράτη-μέλη βλέπουν την επιτακτική ανάγκη να ευθυγραμμίσουν τα προγράμματά τους με τον οικονομικό κύκλο και να θέσουν τις στρατηγικές πολιτικές τους προτεραιότητες τους τομείς αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει σημαντικά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε το ρόλο αυτό στην δημιουργία στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίε θα ψηφιστούν από το Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων του χρόνου τον Ιούνιο. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου. Μία από τις κύριες προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας στα πλαίσια της δημιουργίας μιας ανοιχτής, αξιόπιστης και αναπτυσσόμενης Ευρώπης ήταν η αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Και εκεί αφιερώσαμε ιδιαίτερη προσοχή και χρόνο στην ε, διαμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια ασφαλή πρόσβαση και διέλευση Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση οποιονδήποτε μορφών εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα και πρέπει να συμβάλλει στην ε, γενικότερη εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της πρότασης για το σύστημα φίξεων και αναχωρήσεων. Επομένως, η Ελληνική Προεδρία θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δουλειά βασισμένη στο κείμενο που θα λάβει από εμά. Το Συμβούλιο επίση έχει προχωρήσει στην εξέταση ενό άλλου εγγράφου στα πλαίσια του πακέτου αυτού, του, των καταχωρημένων ταξιδιωτών και του προγράμματο αυτού. Θα μεταβιβάσουμε το θέμα αυτό στην ερχόμενη ελληνική προεδρία. Επίσης, Υπάρχει και ο κανονισμός που ορίζει τις προϋποθέσεις για την διέλευση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων συντονισμένο από την Frontex. Αυτό το εργαλείο πρέπει να είναι αποτελεσματικό ιδιαίτερα όσον αφορά την βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή της Μεσογείου. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι η Προεδρία κατάφερε να οδηγηθεί σε συμφωνία για μια κοινή προσέγγιση στην τελευταία συνεδρίαση της Κοροπέρδη την περασμένη εβδομάδα και ήταν πολύ σημαντικό να ληφθεί η διαπραγματευτική εντολή και με χαρά μου μπορώ να σας ανακοινώσω ότι ήδη διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση σήμερα. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε έναν συμβιβασμό εγκαίρος στο θέμα αυτό. Και εδώ να σας ε, πω ότι για να αποφύγουμε τραγωδίες όπως εκείνη που ζήσαμε πρόσφατα στη Λαμπεντούζα, Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργήσαμε μία task force, μία ομάδα δράσης για τη Μεσόγειο. Όπως ε, συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης-25ης Οκτωβρίου, η Task Force αυτή διεξήγαγε μία διεξοδική ανάλυση της τραγωδίας αυτής και κατέστρωσε ένα σχέδιο δράσης, ένα άμεσο σχέδιο δράσης έτσι ώστε να χειριστεί την κατάσταση και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας θα εγκρίνει το σχέδιο αυτό. Μία άλλη προτεραιότητα της Προεδρίας μας ήταν οι νομοθετικές προσπάθειες για την νόμιμη μετανάστευση. Και εδώ χαίρομαι να σας πω ότι έχουμε καταφέρει να οδηγηθούμε σε ε, θετικά αποτελέσματα για την οδηγία των εποχιακών εργαζομένων. Με την οδηγία αυτή όχι μόνο θα αποφευχθεί η εκμετάλλευση των ε, εργαζομένων αυτών, αλλά θα δοθούν κίνητρα και ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε η προσωρινή διαμονή να μην εξελιχθεί σε μόνιμη διαμονή. Επίσης, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για τις ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές. Ελπίζω αυτό να αποτελέσει μια καλή βάση για την ελληνική προεδρία, έτσι ώστε να συνεχίσει την καλή δουλειά και να οδηγήσει σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Η ψηλά εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την ευρωστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση επίσης ε, για την οδηγία σχετικά με τις έρευνες και τους ερευνητές είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα και ε, συμπεριλαμβάνει πολλούς τομείς της ε, δημόσιας ζωής. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να συνεχίσει η συζήτηση σχετικά με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας αυτής. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας επίσης συνεχίσαμε τις εργασίες μας όσον αφορά τις ε, μεταναστευτικές πιέσεις που ασκούν ορισμένα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο εστίασε τις προσπάθειές τους ε, στους ε, Σύριους πρόσφυγες και στην κατάσταση στη Λαμπεντούσα. Επίσης συνεχίσαμε τους διαλόγους με τις τρίτες χώρες σχετικά με την συνεργασία κινητικότητας με την Ισία, το οποίο και ολοκληρώσαμε και Επίσης υπεγράφει η συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν κατά την ε, διεξαγωγή του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, θα ήθελα να πω ότι με πρωτοβουλία της Λιθουανικής Προεδρίας ενέκρινε τα συμπεράσματά του όσον αφορά τους συναγερμούς. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού 1987-2006 ε, ε, για το δεύτερο, ε, για το σύστημα δεύτερης γενιάς, ΣΥΣ 2 του Σέγγεν. Η εφαρμογή των συμπερασμάτων αυτών θα βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων που φορτώνονται στο σύστημα και θα διασφαλίσει μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών κυρώσεων, περιορίζοντας την κίνηση των επικών τρίτων χωρών στην περιοχή του Σέγγεν. Τώρα, κάνοντας ε, απολογισμό θα ήθελα να αναφερθώ και στο πολύ σημαντικό ε, θέμα της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν ε, για την ε, περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφία των απόψεων στο Συμβούλιο, η Λιθουανική Προεδρία συζήτησε το δεχόμενο να διευρύνει την περιοχή του Σέγγεν, απομακρύνοντας σταδιακά τους ελέγχους στα σύνορα. Δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου όσο πλησίαζε κατέστη σαφές ότι χρειάζεται μια ομόφωνη απόφαση και αυτή δεν καταφέραμε να την έχουμε σε αυτό το στάδιο. Μετά από τις συζητήσεις για το θέμα αυτό και την ε, συμπεριλήφθη και μια κοινή δήλωση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και δηλώθηκε η ετοιμότητα να επιστρέψουμε στην επανεξετάση του θέματος στο μέλλον με σκοπό την επίλυσή του μέσω μιας προσέγγισης σε δύο στάδια. Τώρα, θα ήθελα να προχωρήσω και να σας ε, αναφέρω μερικά ζητήματα όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και της εσωτερικής ασφάλειας. Συζητήθηκε ο κανονισμός Ευρωπόλ, ολοκληρώθηκαν ε, οι διαπραγματεύσεις σε πρώτο στάδιο και έχουμε καταλήξει σε ένα συμβαστικό κείμενο για τα πιο σημαντικά κεφάλαια του κανονισμού αυτού. Το κείμενο αυτό θα υπηρετήσει ως μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Τα περισσοτερα κρατημέλη στο Συμβούλιο εξέφρασαν την άποψή τους και μάλιστα τον Ιούνιο κιόλα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγχώνευση σε πόλη και Ευρωπόλ δεν στηριζόταν σε επαρκή στοιχεία και κάλεσε την Κομισιό να αναθεωρήσει την πρότασή της. Το Συμβούλιο δεν επέστρεψε στο θέμα αυτό και αποφάσισε να μην συζητήσει τους, ε, τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με την συγχώνευση. Ωστόσο, θα ήθελα να πω δύο λόγια παραπάνω για το θέμα σε πόλη και Ευρωπόλ. Όπως ξέρετε, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μην ανανεώσει τη σύμβασή του από, για, τα, για την έδρα της σε πόλη στο Ράμσλι από το 2014. Η Λιθουανική Προεθρία, επομένως, έπρεπε να αντιδράσει γρήγορα και να ψάξει για πιθανές λύσεις που θα διασφαλίσουν την συνέχεια των εργασιών της ΕΣΕΠΟΛ. Το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνη τη 8η ε, Οκτωβρίου κατέληξε σε μια κοινή συμφωνία των κρατών μελών, η οποία έχει ω εξή. Από τη στιγμή που φύγει η έδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή θα μεταφερθεί στην Βουδαπέστη τη Ουγγαρία. Και ε, πληροφορούμε ότι ο Υπουργό Εσωτερικών τη Ουγγαρία χθε παρουσίασε μια εκτενέστατη παρουσίαση για την υποψηφιότητα της ε, Ουγγαρίας και την ε, δυνατότητα μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. 25 κράτη-μέλη υπέβαλαν μία νομοθετική πρωτοβουλία στις 13 Νοεμβρίου, προτείνοντας να τροποποιήσουν το άρθρο 4 της απόφασης ε, του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία της ΕΠΟΛ. Όπως ξέρετε, αυτό το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ειλικρινά ότι η διασφάλιση της συνέχεια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας είναι κοινό μας συμφέρον. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής αυτής, σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Μία άλλη νομοθετική πρόταση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα περισσότερα κράτη-μέλη, είναι η οδηγία PNR για τα δεδομένα των επιβατών. Είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην μάχη κατά της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και διασφαλίζει αποτελεσματική πρόληψη. Επομένω, ένα και περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ε, δρομολογήσει το δικό του σύστημα για δεδομένα των ε, επιβατών και είναι προφανέ ότι χρειαζόμαστε ε, έναν κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίο θα διασφαλίσει την αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία και θα δημιουργήσει επαρκή μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Ελπίζω να λάβετε σοβαρά υπόψη τις δεδομένε συνθήκε προτού αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις για την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία. Τώρα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Το Συμβούλιο συμφώνησε για έναν εποπτικό μηχανισμό και συνοδευτικά μέτρα ασφαλείας. Ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό σε πάνω από μία ευκαιρία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και συζητήσαμε το θέμα και δημερό τους στρατηγικούς μας εταίρους. Στους τομείς της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας ε, τώρα, να σας πω ότι στις αρχές Δεκεμβρίου το Συμβούλιο συζήτησε το ζήτημα των ξένων μαχητών και των όσων επιστρέφουν, ιδιαίτερα στα πλαίσια της εγκατάστασης στη Συρία. Το Συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε ότι ε, πρέπει να εστιάσει τις δράσεις του στον τομέα αυτό, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην δημιουργία ε, καλής ευάσης για ε, δικαστική και ποινική δικαιοσύνη. Και να τονίσω εδώ ότι το Συμβούλιο δήλωσε σαφέστατα ότι για να μπορέσει να εντοπίσει και να ε, ελέγξει το θέμα αυτό των μαχητών χρειάζεται μία ε, αποτελεσματική χρήση του υφιστάμενου συστήματος δεδομένων των επιβατών και μία βελτίωση του μελλοντικού. Και τώρα όσον αφορά το, δεύτε, το, το 2, το ΣΥΣ 2, Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί καλεσμένοι και κυρίες και κύριοι, αυτά είχα να πω και θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ένιωσα μια μεγάλη στήριξη από εσάς. Είχαμε την τύχη να βρεθούμε και στο Βίλνιους με πολλούς από εσάς. Και τώρα θα ήθελα με χαρά μου να ακούσω τα σχόλιά σας και να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Πολλούς βλέπω που θέλουν το λόγο. Συνάδελφοι, έχουμε περίπου μισή ώρα, αν είναι δυνατόν τα σχόλιά σας να είναι σύντομα, ούτως ώστε οι υπουργοί να μπορέσουν να απαντήσουν. Πρώτα θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά θα υπάρξει μια συνολική απάντηση. Πρώτον, κύριε Φλότρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, το πρόγραμμα της CIA για τη μυστική κράτηση είχα μιλήσει στον πρόεδρο στην Ολομέλη από τον Ιούλιο να εκμεταλλευτεί, στην Προεδρόση, στο είχα πει τον Ιούλιο, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ούτω ώστε η Ευρώπη να κάνει ένα βήμα, αποφασιστικό βήμα προς την ασφάλεια, προς την δικαιοσύνη και την αλήθεια για τα προγράμματα, για το ζήτημα αυτό. Ούτε ως χώρο ως Προεδρία αναλάβατε την ευκαιρία αυτή. Μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Πολωνίας γιατί υπήρξε ακρόαση στην Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το ζήτημα αυτό και μάλιστα και εσείς ε, είστε υπόλογοι γιατί έχει γίνει προσφυγή εναντίον σας στη, στο ΕΔΑΔ. Ο πρόεδρος της Πολωνίας είχε πει ότι αν ένας ε, ε υπάλληλος της CIA βασάνιζε κάποιον σε ένα ξενοδοχείο της Βασοβίας θα κατηγορούσε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Αυτό είναι μια προσπάθεια απόσυσης ευθυνών. Έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Δεύτερη ερώτηση. Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας υιοθέτησε μια πρόταση που επιβάλλει, κοινο, που υπο, επιβάλλει κυρώσεις για την ε, άρνηση ηθικών στάσεων και για ανήθικες πράξεις δημοσία. Εμείς αμέσως σκεφτόμαστε ε, ότι αυτό αφορά άτομα που είναι ε, λεσβείες, ομοφιλόφιλοι. Αυτός είναι ο στόχος της νομοθεσίας αυτής. Τώρα, ο συνάδελφος Άλμπρεχτ θεωρεί ότι για τα θέματα της ε, προστασίας δεδομένων δεν έχει προχωρήσει επαρκώς ε, το Συμβούλιο. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης για τις πληροφορίες, να σε ευχαριστήσω για ότι πετύχατε κατά για διάρκεια της και να εκφράσω τη λύπη μου ότι, διότι δεν έγινε δυνατόν να εγκριθεί το πακέτο προστασίας δεδομένων. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι το Κοινοβούλιο έκανε ό,τι μπορούσε ούτω ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής να εγκριθεί το πακέτο προστασίας δεδομένων. Δυστυχώς είχαμε μια πολύ σκληρή θέση του Συμβουλίου στο ζήτημα αυτό. Θέλω να ξέρω γιατί δεν μπόρεσε η Προεδρία σας να προχωρήσει αυτό το πακέτο. Ήταν τόσο σημαντικά. Μίλησε για μητρό επιβατών. Τονίζεται το θέμα των μητρών επιβατών σε μόνιμη βάση. Ωστόσο δεν εγκρίνατε τη δική σας δουλειά, το πακέτο προστασίας δεδομένων. Αν εγκριθεί το πακέτο ε, αν εγκριθεί το μητρό χωρί το πακέτο προστασία δεδομένων θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί υπάρχει λοιπόν το εμπόδιο αυτό. Προ τον Υπουργό Εσωτερικών το πρόγραμμα δράση που δημιουργήσατε με την ομάδα εργασία για την ε, Μεσόγειο και που θα υποβάλλετε συμπεράσματα όπως είπε, είπατε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα δράσης, για την αντιμετώπιση της ε, κρίσεων όπως αυτών που, είχε, που είχαμε στη Λαμπεντούζα. Επίσης, σε τι συνίσταται η συμφωνία κινητικότητας με την Τινησία. Η κυρία Ζήπαλη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Άκουσα τις παρουσιάσεις με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην εισαγωγή του Υπουργού Μπερνατώνης. Άκουσα πάρα πολλά για οικονομία, πολλά για ποινικέ διώξει για θεμελιώδη δικαιώματα και προστασία της δημοκρατίας. Και για να είμαι ειλικρινής, ε, μου έχουν δημιουργηθεί ήδη σκέψεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να εστιάσω στα ακόλουθα σημεία. Καταρχάς ε, αναφέρατε τα εγκλήματα μίσου. και πολύ σωστά το κάνατε. Ε, αναρωτιέμαι όμως ε, και αυτή η ερώτηση απευθύνεται σε εσά ως μέλος του Συμβουλίου και όχι ως πρόεδρο του Συμβουλίου. Αναρωτιέμαι όμως τι γίνεται με τα ακροδεξιά κόμματα. Και τι γίνεται με τις ε, περιπτώσεις των, ε, της ε, μετανάστευσης των Ρωμά και με τις αντιδράσεις των πολιτικών. Σε ορισμένα μέρη, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία παρατηρούμε μάλιστα αποκλεισμό. Όχι θεωρητικό αποκλεισμό αλλά και ουσιαστικό αποκλεισμό. Αποκλεισμό των ε, Ρωμά από την εκπαίδευση, από την αγορά εργασίας. Επίσης, θεωρώ πως πρέπει να εστιάσουμε στο πρόβλημα της διαφθοράς και να συζητήσουμε τα προβλήματα των μειονοτήτων στην Κροατία και σε άλλες χώρες. Τα, ε, οι μειονότητες οι οποίες ε, σημειώνουν σοβαρά προβλήματα. Θα λοιπόν, ε, αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι κάνετε όταν βλέπετε πως οι άλλες χώρες περιορίζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Επίτα, ε, θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο στην απλοποίηση των, των ποινικών διαδικασιών αλλά και από την άλλη όμως πλευρά της δικαιοσύνης, δηλαδή από την πλευρά της υπεράσπισης, εννοώ τα δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας τα έξυπνα σύνορα και ότι αυτά είναι έτοιμα, ότι έχουν επενδυθεί πολλά κονδύλια σε αυτά. Όμως, όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα, ιδιαίτερα για, την, ε, για το ευεργέτημα της ε, παινίας. Πώς αυτό συνδέεται με τις περικοπές που πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει όσο θα έπρεπε. Επίσης, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ληφθούν βιαστικές αποφάσεις και πραγματικά ε, δεν ξέρω τι να πω, διότι πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρο, θα έπρεπε να είναι περισσότερο αναμεμειγμένο στην διαδικασία, να είναι μπροστά από την Κομισιόν και τουλάχιστον να συμπεριλαμβάνεται και το Κοινοβούλιο στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και με πολύ λύπη διαπιστώνω ότι δεν, έχουν, δεν έχει γίνει κάποια νέα συζήτηση, αλλά επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Και γελάνε οι Αμερικάνοι μαζί μας, οι Αμερικανοί φίλοι μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για αυτά που κάνουμε με την ε, προστασία των δεδομένων. Και πιστεύω πως δεν πρέπει να χρονοτριβούμε άλλο, αλλά να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις οι οποίες θα μας προχωρήσουν μπροστά έτσι ώστε επιτέλους να μπορούμε να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική πολιτική για την προστασία των δεδομένων. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην NSA διότι αναφέρατε ε, την Ευρωπαϊκή μνήμη. Όμως, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν είναι οι πράξη των ΗΠΑ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς εμείς στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε και αντιδρούμε ε, με αυτά που μαθαίνουμε πως κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες και πώς εμείς χειριζόμαστε τις μυστικές μας υπηρεσίες. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει κάποια πρόταση, κάποιες ιδέες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πράξεις αυτές των μυστικών υπηρεσιών ή όχι. Το θέμα της προστασίας δεδομένων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων γενικότερα και των δυνατοτήτων που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες, πιστεύω πως συνδέεται άρρηκτα με το κράτος δικαίου και την δημοκρατία στην Ευρώπη και το τι ακριβώς κράτος δικαίου και ποια δημοκρατία θέλουμε και πραγματικά να επαναλάβω ότι ανησυχώ πάρα πολύ με, την, ε, με το δρόμο προς τον οποίο βαδίζουμε. Ωστόσο πρέπει να αναγνωρίσω πως έχετε δώσει κάποια πολύ θετικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αντιπροσωπεύω το ΕΛΚ και είναι μια ομάδα η οποία θεωρεί πως ε, η ασφάλεια είναι ύψης της ε, σημασίας και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και άκουσα σήμερα ότι έχετε καταφέρει να οδηγηθείτε σε έναν καλό συμβασμό με το Συμβούλιο. Όμως ε, πρόσφατα έμαθα κάτι το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ και αφορά την προστασία των δεδομένων και δεν ενοχλεί και δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και πολύ κόσμο. Υπάρχει γενικά γανάκτηση στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση ε, της προστασίας των δεδομένων και το τι γίνεται με την Αμερική, ιδιαίτερα από τότε που έγιναν οι αποκαλύψεις από τον Edward, Edward Snowden για την κατασκοπία των Ευρωπαίων πολιτών από, την, ε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρχισαν να αυξάνονται και οι πιέσεις προς τα εμάς για ε, επικύρωση τη ε, συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, η Επίτροπο Ρέντινγκ είχε υποστεί πάρα πολλές πιέσει. όμως το θέμα τη ε, της των δεδομένων παραμένει και γι' αυτό μπήκαν στον πάγο οι διαπραγματεύσεις και εμείς πιστεύω ότι με αφορμή αυτό και με αφορμή την, τις που δημιουργήθηκαν στη συνείδηση των Αμερικανών. Έχουμε πλέον ένα ανοιχτό παράθυρο ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε. Και πιστεύω πως η Επίτροπος Ρέντιν κατάφερε να κάνει καλή δουλειά στις διαπραγματεύσεις και όμως υπάρχουν, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και τα κράτη-μέλη είναι διχασμένα όσον αφορά την στάση τους προς τη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ να πω ότι ενοχλούμε και ως Ευρωπαίος και ως Ευρωβουλευτής για το ότι υπάρχουν διχασμένες ε, απόψεις και στάσεις σχετικά με τις ε, σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή θέση και γι' αυτό θα παρακαλούσα να το λάβει υπόψη του το Συμβούλιο αυτό στις μελλοντικές του διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μάλλον ε, αναφέρθηκε στα εγκλήματα ε, μίσους ο Υπουργός Περνατώνη. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχουν αναγνωριστεί οι ειδικέ κατηγορίες με βάση την εθνοτική προέλευση, γενετήσιο προσανατολισμό ε, ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο κριτήριο. Έχετε λάβει υπόψη να μιλήσετε για μια ενιαία ενιολογική βάση για το μίσος, για εγκλήματα μάλλον μίσους, τη στιγμή που ε, βασίζονται αυτά τα εγκλήματα σε, ε, στην ιδεολογία ή σε πολιτικές προτιμήσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στον ενιαίο κατάλογο για εγκλήματα μίσους. Θα ήθελα, λέει ο Πρόεδρος, να υποβάλω κι εγώ μία ερώτηση. Σταθήκατε στο θέμα του Ευρωπαϊκού PNR. Με βάση την παρούσα θέση μας και την πρόοδο στη Γαλλία με το δικό της σύστημα, καθώς και τη χρηματοδότηση ε, σε άλλα 12 κράτη-μέλη, υπάρχουν μεγαλύτερες ανησυχίες, ιδιαίτερα με τους ξένους, τους αλλοδαπούς μαχητές και το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θεωρείτε ότι το ευρωπαϊκό PNR θα μπορούσε να είναι προτεραιότητα για το μέλλον και θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ε, αυτή είναι η δική μου ερώτηση, αλλά έχετε πληθώρα ερωτήσεων να απαντήσετε. Δεν ξέρω ποιος θα αρχίσει. Έχετε το λόγο. Ο κύριος μάλλον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ε, πράγματι, Πρόκειται για σωρία ερωτήσεων και όλες είναι σχετικές με το χαρτοφυλάκιό μου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Η ερώτηση της κυρίας Φλότρ για τα κέντρα κράτησης. Θεωρούμε ότι κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δηλαδή, εάν υπάρχουν τέτοιοι ισχυρισμοί θα πρέπει να διερευνηθούν. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση κάποια τεκμηρίωση. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη φέρουν ευθύνη με βάση το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. Η Λιθουανική Προεδρία θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα. Και αυτό το ε, ανέφεραν και οι Υπουργοί Εσωτερικών. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να αναλάβει δράση πάντα, αλλά ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τις διατάξεις των ε, διεθνών συνθήκων και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των προσφύγων. Η Λιθουανία είναι το μόνο κράτος που διενέργησε διεξοδικές διερευνήσεις και προέβησε έρευνες για τη μεταφορά προσώπων σε αυτά τα κέντρα κράτησης και δεν, τουλάχιστον στη Λιθουανία, στο δικό μας έδαφος, δεν υπήρχαν τέτοια παράνομα κέντρα κράτησης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την ύπαρξή τους χωρίς τεκμηρίωση. Ως προς τις διοικητικές κυρώσεις που προευλήθησαν, Νομίζω ότι το θέμα σχετίζεται με τη χώρα μας και την Προεδρία. Σε σχέση με τις διοικητικές κυρώσεις κατά τον ΛΟΑΔ, θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τύχει προτεραιότητας. Στο πρόγραμμα της Προεδρίας μας ανέφερα το γεγονός, αναφέρθηκα στο γεγονός ότι δεν προβλεπόταν μία ειδική σύσκεψη για τους ΛΟΑΔ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης πάντα υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ και εάν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Εγώ ως Υπουργός δεν ε, δέχομαι αυτές τις, ε, ε, αυτές τις αιτιάσεις. στην ομάδα εργασίας ασχοληθήκαμε επί 20 μέρες για το θέμα. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο και κατά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών στο Βίλνιους. Όμως το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου προβλήθηκαν νέες νομικές πτυχές επί του θέματος και η νομική υπηρεσία προέβαλε αυτά τα ζητήματα. Τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να λάβουν αποφάσεις γιατί δεν υπήρχε εξισορρόπηση μεταξύ ε, των συμφερόντων ε, των επιχειρήσεων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δέχομαι λοιπόν αυτά που είπαν τα μέλη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό δεν ελήφθηκε απόφαση το Δεκέμβριο, διότι μερικοί υπουργοί δεν ήταν απόλυτα σίγουροι για την εμφέλεια του ζητήματος. Πιστεύω ότι οι συζητήσεις περί προστασίας δεδομένων προβάλλουν ένα εύρος δυνατοτήτων. Και ο Υπουργός της Ελλάδας είναι της ίδιας γνώμης. Ίσως θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στην αρχική πρόταση. Πιστεύω όμως ότι αυτή είναι η προσέγγιση του ζητήματος και από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ως προς την ε, προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το Συμβούλιο προσέδωσε μεγάλη σημασία στο ζήτημα Εάν ε, συμμετείχατε στη διάσκεψη του Βιλνιούς θα το διαπιστώσατε αυτό. Ε, διοργανώθηκε αυτή η συνάντηση από τη Λιθουανική Προεδρία μαζί με τον Οργανισμό ε, Υπεράσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συζητήσαμε και για εγκλήματα μίσους που σχετίζονται με τους Ρωμά ε, καθώς και σεξουαλικές μειονότητες. Η διάσκεψη, η διάσκεψη κρίθηκε θετικά και το Συμβούλιο το Δεκέμβριο ενέκρινε την έκθεση για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάσαμε σε συμπεράσματα σε σχέση με την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους και φτάσαμε σε μια κοινή θέση. Άρα δεν συμφωνώ με τη γνώμη σας ότι δεν επετεύχθη τίποτα. Πάντα είμαι ε, έτοιμος να δώσω περαιτέρω πληροφορίες εάν δεν ε, τις διαθέτετε επί του θέματος. Ε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ο Υπουργός Μπαρακάουσκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω. Η κυρία Ρομέρο υπέβαλε ένα ερώτημα και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ως προς την ε, ευρωπαϊκή δράση στη Μεσόγειο, ζήσαμε μια μεγάλη τραγωδία, αναμφίβολα, και με ρωτήσατε ποια ήταν τα συμπεράσματα της Task Force για τη Μεσόγειο, καθώς και τη γνώμη μου για το κατά πόσο τα προτινόμενα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκούν για να προλάβουμε μια άλλη τραγωδία. Όπως γνωρίζετε, η Task Force για τη Μεσόγειο που συστάθηκε μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προέβη στην ανάλυση της κατάστασης και αποφάσισε να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο και τη βελτίωση της κατάστασης. Η Task Force ήδη συνήλθε δύο φορές και τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων δημοσιεύτηκαν στο ανακοινωθέν τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ανακοινωθέν αυτό υπευλήθη στη συνέχεια στο Συμβούλιο και κρίθηκε πολύ επικοδομητικό και επίκαιρο. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι ο μηχανισμός διάσωσης στη θάλασσα θα πρέπει να ενισχυθεί, να είναι πιο αποτελεσματικός. Επίσης, το Συμβούλιο τόνισε το γεγονός ότι χρειάζεται συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν πρέπει να αναλαμβάνεται μεμονωμένα από τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με την αντιμετώπιση τρίτων χωρών στην ε, Μεσόγειο. Επίσης αποφασίστηκε να δράσει η Frontex καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τους Πρόσφυγες. Θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως και ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες προέλευσης ή διαμετακόμισης. Θα πρέπει να προωθηθεί αλληλεγγύη με αυτές τις χώρες, όπου βεβαίως υπάρχουν πιο έντονες μεταναστευτικές ροές. Επίσης η Europol θα πρέπει να δράσει αμεσότερα, ιδίως άμα πρόκειται, άμα έχουμε να κάνουμε για, ε, με παράνομο εμπόριο, μετανάστευση και οργανωμένο έγκλημα. Προσπάθησα να σας απαριθμίσω τις θέσεις του Συμβουλίου και το τι επιτύχαμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ναι, ναι. Είχα και εγώ ερωτήσεις από την Πρόεδρο. Είναι αυτονόητο, Πρόεδρε, ότι το εργαλείο αυτό είναι ενδιαφέρον για μας. Η Προεδρία λοιπόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και με χαρά ακούσαμε ότι η απόφαση ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να ασχολείται με την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Πιενάριο σύλλεξαμε όλες τις πληροφορίες από τις χώρες τις οποίες ε, υπάρχουν ε, PNR ε, συστήματα και καταφέραμε να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριοι Υπουργοί, όχι μόνο και για την συνολική παρουσίασή σας, αλλά και γιατί απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Θέλω να σε ευχαριστήσω και για τη δουλειά που κάνατε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τον καινούργιο χρόνο, καθώς και καλά Χριστούγεννα για σας και για τον λαό της Λιθουανίας συνολικά. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι στη φάση αυτή θα μπορούσα να διακόψω, αν να προσθέσω απλά δεν έχω κάτι άλλο. Η επόμενη συνάντηση Έχουμε βέβαια και άλλο θέμα στις 5. Έρευνα της Επιτροπής ΒΥΜΕ για την ηλεκτρονική μαζική επιτήρηση πολιτών της Ένωσης. Και αύριο θα τα πούμε στις 9 στο 2Q2. Διακόπτουμε τώρα μέχρι τις 5. Thank you very much. <laughs> Uh, Κινούμε, συνάδελφοι. Συγγνώμη που καθυστερούμε και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Συγγνώμη και ξανά για την καθυστέρηση η παρουσίαση του εγγράφου εργασία για την ε, Ευρωπαϊκή και Εθνική Ασφάλεια από την οπτική γωνία της Ένωσης θα καθυστερήσει. Δεν θα γίνει αύριο στις 11. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, να εγκρίνουμε την υπόλοιπη μερίσια διάταξη για σήμερα και αύριο. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν μαλτέζικα και δεν υπάρχουν φιλανδικά. Συγγνώμη γι' αυτό. Κροατικά, συγγνώμη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διάσκεψη και συγγνώμη από τους συναδέλφους που περίμεναν με υπομονή στην άλλη πλευρά. Θα μιλήσει η κυρία Βανέσα την πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έρευνα για την κατασκοπία και τον κύριο Ρικάρντο Ρεζέντε, εισηγητή τη κοινοβουλευτική ε, Εξεταστική επιτροπή για την κατασκοπία. Α του ακούσουμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσετε εισαγωγικά, να σας τονίσω θα ακούσουμε και τους δύο συναδέλφους από την γερουσία της Βαζιλίας μετά την ε, ε, πληροφορία ότι υπήρξε παρακολούθηση της Προέδρου της Βραζιλίας, υπουργών αλλά και επιχειρηματιών. Ξεκίνησε μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή από την γερουσία της Βαζιλίας για το θέμα αυτό που συναντήθηκε ε, που επικοινώνησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2013 με εμά για να ζητήσει τις δικές μας απόψεις. Ο πρόεδρος Σούλτς και εγώ στείλαμε επιστολή στον πρόεδρο της Γερουσίας και της Επιτροπής σχετικά και σήμερα θα ακούσουμε εν τέλει με βίντεο διάσκεψη την κυρία Γκρατσιωτίν, πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και τον εισηγητή κύριο Ντερεζέντε Φεράσο. Σας ευχαριστώ που συναντιόμαστε. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Κυρία Γκρατσιωτίν, έχετε το λόγο, αλλά δεν είναι εδώ η κυρία Γκρατσιωτίν, αλλά έχουμε τον κύριο Ρικάντο Τριζέντε Φεράσο. Ε, έχετε το λόγο. Relator da Comissão de Investigação no Senado brasileiro. Η εξεταστική των πραγμάτων ε, επιτροπή που συστάθηκε στη Βραζιλία θα ήθελε να σας ενημερώσει. Η κυρία Βανέσα Γκρατζιωτίν είναι η πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής και καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας έδωσε ο Ευρωβουλευτής Κλάουδιο Μωράης και οι συνάδελφοί του, διότι με αυτή την ανταλλαγή απόψεων μπορούμε να φτάσουμε σε κοινά συμπεράσματα. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια της χώρας μου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθώντας να τελειοποιήσουμε, να ερευνήσουμε ε, τρόπους και μέσα έτσι ώστε τα κράτη μας να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό μαζί με τους συμπατριώτες μας, έτσι ώστε να δώσουμε στους συμπατριώτες μας τη δυνατότητα να νιώσουν πιο ασφαλείς στον ιδιωτικό τους χώρο. Αυτό αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τις επιχειρήσεις. Διαθέτουμε πληροφορίες για ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τις χώρες μας. Βεβαίως καταληφθήκαμε εξαπίνης όταν μάθαμε για τις υποκλοπές και την κατασκοπία που αποκάλυψε ο Έντουαρτ Σνόουντεν. Θελήσαμε λοιπόν να επαληθεύσουμε τα πεπραγμένα. Έγιναν πολλές ακροάσεις που όρισε, όρισαν οι εκτελεστικές αρχές. Ανελήφθησαν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε κοινέ δημόσιες πολιτικές, μια δημόσια πολιτική για να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ορίζοντας μία εθνική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της παραβίασης του κυβερνοχώρου και της ιδιωτικής ζωής. Το Δεκέμβριο θα καταλήξουν οι εργασίες μας τον Δεκέμβριο του 2013. Κρίναμε όμως ότι θα ήταν σκόπιμο να παρατείνουμε αυτή την προθεσμία έτσι ώστε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προωθήσουμε αυτό το διάλογο, αυτές τις επαφές, έτσι ώστε να δράσουμε από κοινού. για να προβούμε σε κοινέ στοχοθετήσεις. Πρόκειται για παραβιάσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την... και ε, αναγνωρίστηκαν ιδιαίτερα από την NSA. Εμείς θέλουμε να προβούμε σε αυτή την επικοδομητική συνεργασία και αντιμετώπιση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να οριοθετήσουμε τα πράγματα στις παραβιάσεις αυτές οι οποίες είχαν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας από τον Έντουαρτ Snowden. Δίλμα Ρουσέφ, όπως ξέρετε, κατήγγειλε το γεγονός ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, υπερασπιζόμενη τον βραζιλιάνικο λαό. Προσπαθούμε λοιπόν να ορίσουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια της κυβέρνησης και μέτρα που θα μπορέσουμε να λάβουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την προστασία και των, των πολιτών και να προστατεύσουμε γενικότερα τον ιδιωτικό τους βίο. Πρόκειται για πληροφορίες στρατηγικής σημασίας. Η τηλεδιάσκεψη αυτή έχει μεγάλη σκοπιμότητα μέσα στα πλαίσια της ε, συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να συγκλίνουν οι απόψεις μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε μια κοινή δράση. Στις αρχές ε, του Φεβρουαρίου θα μπορέσουμε να συναντηθούμε. Θα συμμετέχει και η κυρία Βανέσα Γκραζιωτίν θα προτείνουμε λοιπόν μια νέα τηλεδιάσκεψη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα συμπεράσματα της εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. έτσι ώστε να προβάλλουμε μια κοινή αντίδραση και αντιμετώπιση. Θα θέλαμε η πρότασή μας να αποτελέσει έναν έναυσμα συνεργασίας με την περιοχή του Μερκοσούρ. Έτσι ώστε Μερκοσούρ και Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσουν ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μέσα στα πλαίσια μιας συμφωνίας, γενικότερης συμφωνίας που προωθούμε εδώ και χρόνια. Θα προβάλλουμε δηλαδή το αίτημα μια κοινή συνάντηση είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε εδώ στη Βραζιλία έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτά είναι τα λόγια τα λίγα λόγια εισαγωγής από δικής μου πλευράς και θα ήθελα και τις δικές σας απόψεις ε, ως προς τη διερεύνηση αυτή. Ο Έντουαρτ Σνόντεν δημοσίευσε σε μια μεγάλη εφημερίδα του Σάου Πάουλο μια ανοιχτή επιστολή προς τον βραζιλιάνικο λαό, που εκδηλώνει την, ε, δηλώνει μάλλον την ικανοποίησή του, διότι η Βραζιλία ε, αντέδρασε τόσο άμεσα στις καταγγελίες αυτές. Και ζήτησε τη συνεργασία με γερουσιαστές της ε, γερουσίας της Βραζιλίας επί του θέματος. θεωρεί ότι η θέση του είναι επισφαλή στη Ρωσία, όπου έχει ζητήσει και ε, πολιτικό άσυλο και ενδεχομένως ζητήσει πολιτικό άσυλο και από τη δική μας χώρα έτσι ώστε να μπορέσει να συνεργαστεί στη διερεύνηση αυτών των καταγγελιών. Να μπορέσει να συνεργαστεί μαζί μας στα πλαίσια της ε, διαλεύκανσης του όλου πλαισίου παραβίασης του κυβερνοχώρου και της ιδιωτικής ζωής. Έτσι ώστε να ε, αντιδράσουμε συλλογικά. Η πρόεδρος της Δημοκρασίας της Δημοκρατίας μπορεί να χορηγήσει άσυλο, αλλά και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη, της Γερουσίας υποστήριξε την κυβέρνηση της Βραζιλίας θεωρώντας ότι θα πρέπει να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στον κύριο Σνόουντεν εδώ στη Βραζιλία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε εκ του σύνεγγης και να διερευνήσουμε αυτές τις ε, καταγγελίες. Θα δώσω το λόγο στην ε, πρόεδρό μας, την κυρία Βανέσα Γκραζιοτσίν, η οποία συντονίζει τις εργασίες μας και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η κοινή προσπάθεια είναι ύψης της σημασίας μέσα στα πλαίσια της αποφασιστικότητάς μας να αντιμετωπίσουμε από κοινού το ζήτημα αυτό. Να υπάρξει δηλαδή μια κοινή αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της Βραζιλίας για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε καλύτερα στα πλαίσια αυτών των συνεχών παραβιάσεων. Θα δώσω το λόγο τώρα στην γερουσιαστή Βανέσα Γκραζιοτσίν που είναι πρόεδρος της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής. Ελπίζω το Φεβρουάριο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μέσα στα πλαίσια μίας ε, κοινή συνεδρίασης, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε εδώ στη Βραζιλία, με τη δική σας συνεισφορά κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ορίζοντας ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε συνεργασία και με το Μερκοσούρ. Η κυρία Γκραζιοτσίν έχει το λόγο. Καλό σας απόγευμα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αποτείνω ένα χαιρετισμό και από πλευράς των συνεργατών, γερουσιαστών και του εισηγητή του γερουσιαστή Ρικάρντο Φεράσου που ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό εκ του σύνεγγης μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της Γερουσίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την τεκμηρίωση που μας αποστήλατε και θα μας αποστήλετε και στο μέλλον. Θεωρούμε λοιπόν με βάση και τη δική μας ε, τεκμηρίωση ότι έχουμε να κάνουμε με κοινούς ε, στόχους. Διαβάζοντας τα δικά σας έγγραφα μπορώ να τονίσω ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί και οι εργασίες μας. Έχει βεβαίως σημασία και η συνεργασία στον, στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο επιχειρήσεων. Εσείς είσαστε πολύ πιο προηγμένοι σε αυτό το τομέα. Μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο των υποκλοπών και της κατασκοπίας που αφορά φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και δυστυχώς και η πρόεδρός μας, η Ντίλμα, αποτέλεσε αντικείμενο αυτής της κατάφορης παραβίασης, δηλαδή έγινε υποκλοπή στο κινητό της τηλέφωνο, κάτι το οποίο κατήγγειλε και η ίδια. Άρα η κατασκοπία έγινε και σε κρατικό επίπεδο και σε επίπεδο ανώτατων αξιωματούχων. Άρα θα πρέπει να προβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις με βάση αυτές τις καταγγελίες για την ε, παραβίαση του ιδιωτικού βίου αλλά και του δημοσίου. Ο εισηγητής μας, ο, ο Ρικάρντο Ντερεζέντε Φεράσου, θα προβεί και σε μία δημοσίευση. Δεν ξέρω ε, κατά πόσο σας μίλησε ο κύριος Φεράσο για την ενδεχόμενη χορήγηση πολιτικού ασύλου προς τον κύριο Σνόντεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί. Δεν μπορούμε εμείς να ασχοληθούμε άμεσα με αυτό το αίτημα και δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του αιτήματο του κυρίου Σνόουντεν και της, ε, των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά διαβήματα δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, ούτε μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα σχήμα ανταλλαγών. Δηλαδή, αν του χορηγήσουμε άσυλο, τότε θα προωθηθούν και οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα πρώτα βήματα διαλόγου, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και το Φεβρουάριο και η κυβέρνηση της Βραζιλίας θα διοργανώσει μία διάσκεψη τον Απρίλιο του 2014 σε παγκόσμιο επίπεδο για τις ε, καταγγελίες των κυβερνοχώρο. Ο πρόεδρος Ολάντ βρέθηκε στη χώρα μας και με την πρόεδρό μας, τη Ντίλμα Ρουσέφ, τόνισε ότι θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η διεθνής διάσκεψη για τις παραβιάσεις και καταγγελίες στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να προβάλλουμε ένα ε, δημοκρατικό διαδίκτυο όπου όμως δεν θα παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ιδιωτικού ε, βίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ανταποκριθήκατε άμεσα. Χαίρομαι που διοργανώθηκε αυτή η τηλεδιάσκεψη στο Βραζιλιάνικο Κογκρέσο έχουμε πολλές εργασίες, θα ψηφίσουμε και τον προϋπολογισμό το Φεβρουάριο όμως θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις εργασίες ίσως εκ του σύνεγγης. Θα ήθελα να ε, τονίσω προς τον Κλάουντιο Μωράης ότι το 2001 το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε ε, με μία διερεύνηση των υποκλοπών, των τότε υποκλοπών. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς αξιολογήσατε την κατάσταση διαχρονικά. Ποιες είναι οι διαφορές με αυτή τη νέα συγκυρία που ζούμε σήμερα. Okay, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο κυρία και κυρία Τερέζαν Τεφεράς, Ελπίζω να πρόφερα τα όνοματά σας σωστά. Μπορείτε να με ακούσετε καλά, διότι είχατε πει προηγουμένως ότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Μπορείτε να με ακούσετε καλά. Ναι. Πολύ καλά. Ε, μην θεωρήσετε δεδομένου ότι μιλώ πορτογαλικά επειδή έχω πορτογαλικό επώνυμο. Ε, μπορώ να καταλάβω λίγα πορτογαλικά. Καταρχάς ε, είστε στη θέση εισηγήτριας διότι μου κάνετε ερωτήσεις αλλά εμείς είμαστε εκείνοι που για το εσελόν αλλά εμείς είμαστε αυτοί που θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για την σημαντική συνεισφορά σας. Είναι προφανές ήδη ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων ανάμεσα στη δική σας ε, Διερευνητική Επιτροπή και εμάς. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Γι' αυτό να πω ότι καταρχάς είναι πολύ θετικό ε, το ότι δηλώσατε πρόθυμοι να γίνει μια συνεδρίαση, μια συνάντηση το Φεβρουάριο και εμείς έχουμε πολλά πράγματα στο πρόγραμμά μας όπως και εσείς, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να συναντηθούμε τον Φεβρουάριο και να ανταλλάξουμε πληροφορίε. Είμαι πρόεδρο εδώ σε αυτή τη συνεδρία, είμαι όμω και εισηγητή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σα πω κάποια πράγματα για το Ισελαιόν και για το τι έγινε το 2010. Ένα από τα ε, σημαντικά σημεία ήταν ότι οι συστάσεις του Ισελαιόν δεν εφαρμόστηκαν. Η έκθεση αυτή ήταν εξαιρετική και ελπίζω τον Φεβρουάριο κάποια από τα στοιχεία αυτά, κάποιες από τις συστάσεις να συμπεριληφθούν. Καταρχάς, αντί εισαγωγής θα ήθελα να ε, σας ρωτήσω δύο πράγματα και πιστεύω πως έχουμε αρκετό χρόνο για να συγκεντρώσουμε ερωτήσεις, τρεις ίσως και να τις απαντήσετε μαζί. Τρεις ερωτήσεις κάθε φορά οι δικές μου ερωτήσεις. Πρώτον, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες ε, στις δύο επιτροπές, τη δική σας και τη δική μας και τις έρευνές μας, θα ήθελα να σας ερωτήσω ε, ε βασισμένο στα στοιχεία που μας παρουσιάσατε, το εξής. Είχαμε πολλές ε, συνεδριάσεις διερευνητικών επιτροπών μέχρι τώρα και πιστεύω πως έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να έχουν δυνατότητες, τις δυνατότητες προσφυγής που θα έπρεπε να είχαν απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και εσείς έχετε ζητήσει μια τέτοια προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς καταλαβαίνετε εσείς τις εξελίξεις και την πρόοδο των ερευνών σας. Τι πιστεύει ο λαός της Βραζιλίας όσον αφορά τις ε, δυνατότητες προσφυγής απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Πώς δηλαδή θα δικαιωθούν οι πολίτες, οι μη Αμερικανοί πολίτες. Έπειτα, όσον αφορά το ψήφισμα πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για, την, ε, για το διαδίκτυο. Ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε δει και από εμάς μεγάλο ενδιαφέρον, από τη Γερμανία ιδιαίτερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω προς τα πού πηγαίνει το θέμα αυτό και ποιες είναι οι επιπτώσεις και για την Βραζιλία και επίσης το πώς ε, αντιμετωπίζετε εσείς το ζήτημα αυτό στις ε, δικές σας έρευνες. Αυτά ε, από εμένα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Άννα Γκόμες για τη δική της ερώτηση και μην ανησυχείτε. Δεν θα κατακλειστείτε από ερωτήσεις Πορτογάλων Ευρωβουλευτών. Όμως τώρα θα δώσω το λόγο στην Άννα Γκόμες, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, καλό σας απόγευμα, συνάδελφοι. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής της Γερουσίας, θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα ορίσετε ε, την προσφυγή στη δικαιοσύνη, judicial redress. Διότι σύμφωνα με τον νόμο των ΙΠΑ, ένας αλλοδαπός πολίτης δεν μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη μέσα στα πλαίσια ε, ενός δόλιου ε, χειρισμού ή αντιμετώπιση, δηλαδή στα πλαίσια της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας. Εμείς δίνουμε μεγάλη μάχη και μέσα στα πλαίσια του Αμερικανικού Κογκρέσου, διότι αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας, η δυνατότητα προσφυγής για να οικοδομηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προστασίας δεδομένων που να αντικατοπτρίζει τα πρότυπά μας ως προς την ε, υπεράσπιση του ιδιωτικού βίου και την προστασία δεδομένων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε τους Αμερικανούς για κάτι τέτοιο. Ακόμα και στις σημερινές μας επαφές με μία αντιπροσωπεία του Κογκρέσου υπό τον Μάικ Ρότζερς είδαμε ότι δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης του ζητήματος. Πώς κινείστε εσείς σε αυτόν το τομέα, προβάλλετε παρόμοιες απαιτήσει στους Αμερικανούς. Πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στη συνεργασία που έχετε με τους Αμερικανούς ως προς την μεταβίβαση ε, προσωπικών δεδομένων, ε, τα προγράμματα PNR, δηλαδή τον κατάλογο επιβατών που απαιτείται από τις αεροπορικές μας εταιρείες και από τις δικές σας. Σε αυτό το τομέα νομίζω ότι σίγουρα θα μπορούσαμε να προβάλλουμε ένα κοινό μέτωπο και αυτό προς ε, κοινό συμφέρον. Τρίτη ερώτηση από την κυρία Σίπελ, Γερμανό, Γερμανίδα από την Επιτροπή Λίμπε. Ελπίζω να... Η ερώτησή μου να είναι καλή. Καταρχάς, Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα για αυτήν την ε, βιντεοδιάσκεψη, διότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθούμε τις συζητήσεις μετά από τις αποκαλύψεις του Edward Snowden, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες και σε εσάς. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι ευπρόσδεκτη η συνεργασία. Αν κατάλαβα καλά, στην Βραζιλία έχουμε μια παρόμοια κατάσταση με εδώ. Έχετε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες σας στην Διερευνητική Επιτροπή. Όμως θα ήθελα να ξέρω θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι τομεί στους οποίους πιστεύετε ότι πρέπει να εργαστείτε περισσότερο έτσι ώστε να καταλήξετε σε συμπεράσματα. Χρειάζονται καινούργιοι νόμοι, καινούργιοι κανόνες σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ε, πιστεύετε πως χρειάζονται τεχνικές λύσεις έτσι ώστε το διαδίκτυο να γίνει ασφαλέστερο ε, και να προστατεύει καλύτερα την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα των χρηστών. Τέλος, ε, υπάρχουν κάποιες ιδέες για νέους κανόνες που θα διέπουν τις μυστικές υπηρεσίες τι, κάποιες εξουσίες που οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό. Ε, να πω τέλος ότι παρότι ενδεχομένως να υπάρχουν μικρές διαφορές από χώρα σε χώρα, να ανάμεσα σε εσάς και εμάς, ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα και κοινά μέτρα διότι παρότι βρισκόμαστε σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, σκεφτόμαστε όλοι για τα ίδια πράγματα, για τα ίδια θέματα και θέλουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως θα βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει όλο αυτό ταυτόχρονα από κοινού. Τέλος, κάτι που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξή. Αναφέρατε την επιστολή του κυρίου Σνόντεν προς τον λαό της Βραζιλίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι αντιδράσεις του κοινού του λαού της Βραζιλίας σε αυτή την επιστολή. Επίσης, καταστήσατε σαφές ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ίδια την ε, έρευνα που διεξάγεται και στο θέμα του ασύλου. Όμως ε, συζητείτε το θέμα αυτό και εδώ στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν θα σας ρωτήσω αν θα δώσετε άσυλο στον Edward Snowden, διότι πιστεύω πως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις, αλλά πιστεύετε ότι μόνο και μόνο από τις αποκαλύψεις του κυρίου Snowden έχει δοθεί δυνατότητα για να γίνει αυτή η συζήτηση και γι' αυτό και εσείς και εμείς και άλλα μέρη στον κόσμο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς θα δώσουμε άσυλο ή προστασία στον κύριο Σνόντεν. Θα ήθελα να επιστρέψω τώρα, λέει ο πρόεδρο, στου συναδέλφου από τη Βραζιλία, να του ζητήσω να απαντήσουν στι ερωτήσει αυτέ και να του ζητήσω κατά την απάντησή του να μα ε, δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες, διότι και μας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμείς βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης της έκθεσης και γι' αυτό θα μας, ε, ε, ενδιαφέρει πολύ η απάντησή σας. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να αρχίσω. Ο γερουσιαστής Ρικάρντο Φεράσου μίλησε πολύ περισσότερο από μένα κατά την εισήγησή του. Εγώ θα απαντήσω στις επιμέρους ερωτήσεις. Θα αρχίσω από την τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δόθηκε να απαντήσουμε. Ως προς το αίτημα του κυρίου ε, Σνόντεν, η επιστολή ε, ελήφθη, παρελήφθη εχθές. Είναι κάτι το πολύ πρόσφατο και το είδε ο πολύς ο κόσμος στο διαδίκτυο και στον τύπο σήμερα. Δεν έχουμε ε, πολλά νέα ως προς τις αντιδράσεις του βραζιλιάνικου λαού. Βεβαίως υπήρξαν αντιδράσεις ήδη, μερικοί αντιτάχθηκαν, μερικοί βουλευτές αντιτάχθηκαν στη χορήγηση ασύλου προβάλλοντας το ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μια γενικότερη πολιτική ανησυχία και κλειδονισμούς ενδεχομένως. Άλλοι βουλευτές θεωρήσαν ότι θα πρέπει να χορηγηθεί άσυλο αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που προευλήθη είναι ότι δεν, ε, δεν πρόκειται για έναν κοινό υπόδικο. Ε, δεν έχει προβεί σε κάποιο αδίκημα ή εγκληματική ενέργεια. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις, το φάσμα αντιδράσεων. Θα δούμε ποια θα είναι η τάση που θα διαμορφωθεί στο εγγύς μέλλον. Τώρα, κατά πόσο θα χορηγηθεί ή όχι άσυλο, αυτό αφορά την εκτελεστική αρχή. Εμείς μπορούμε να κάνουμε υποδείξεις αποκλειστικά, να ταχθούμε υπέρ ή όχι, αλλά η κυβέρνηση θα αποφανθεί. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να χορηγηθεί ε, άσυλο στον κύριο Σνόουντεν, διότι θεωρούμε ότι η δράση του ήταν ευεργετική υπέρ όλων των λαών. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ολοένα και διονγκούμενη κατασκοπία αλλά δυστυχώς σύμμαχοι και φίλοι αποτέλεσαν αντικείμενο ε, αυτής της κατασκοπίας. Κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα ατυχές. Σε ποιους τομείς θα ε, συνεργαστούμε. Υπάρχει το διεθνές σκέλος που αφορά την ε, διεθνή κοινότητα και το τοπικό επίπεδο ή κρατικό. Πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα δράσουμε εδώ στη Βραζιλία. Ως προς τη διεθνή αντίδραση, η Βραζιλία γνωμοδότησε σε σχέση με το γεγονός ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία που διέπει το διαδίκτυο ανά τον κόσμο, ακόμα και πριν από τις καταγγελίες του Σνόντεν, διότι η νομοθεσία είναι πολύ χαλαρή και θα πρέπει να είναι πολυμερής και πολυεπίπεδη. Όπως ξέρετε, μαζί με την Γερμανία προβάλαμε ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και προβάλαμε και την Διεθνή Διάσκεψη του Απριλίου που αποτελεί ένα πολιτικό έναυσμα για να αντιδράσουμε όλοι άμεσα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι δυναμικά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δική του πλευρά θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διάσκεψη ύψη της ε, σημασίας τον ε, Απρίλιο. Όσον αφορά τα εσωτερικά ζητήματα της ε, Βραζιλίας, ήδη εγκρίνονται ορισμένα μέτρα το Κογκρέσο. Δηλαδή η Γερουσία και η Βουλή ενέκριναν ένα νομοθέτημα για την ε, κοινή αντιμετώπιση της ε, κατασκοπίας και των ε, υποκλοπών. Επίσης, θα υποβάλουμε και άλλα σχέδια νόμου που θα σχετίζονται με την προστασία του πολίτη γιατί επειδή οι επιχειρήσεις του διαδικτύου είναι κατά κύριο λόγο αμερικανικές, θεωρούν ότι η μόνη δικαιοδοσία είναι εκείνη των ΙΠΑ αλλά ε, ε και οι υπόδικοι σε αυτή την περίπτωση αρνούνται να λογοδοτήσουν ή να δικαστούν από την ε, βραζιλιάνικη δικαιοσύνη. Εμείς θα ζητήσουμε να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα, ως προς την προστασία των δεδομένων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι υπόλογες οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν δραστηριότητα στο δικό μας έδαφος, στη δική μας επικράτεια. Και η Βουλή των Αντιπροσώπων συντάσσει ένα νέο νόμο για την δράση στο διαδίκτυο που θα έρθει στη συνέχεια στη Γερουσία. Υπάρχει και ένα ε, μείζον ζήτημα, διότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο δράσης των επιχειρήσεων διαδικτύου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα data center εδώ στη Βραζιλία. Αυτό αφορά ε, θέματα ασφάλειας, ασφάλειας των πολιτών σε σχέση δηλαδή, σχετίζεται δηλαδή με την προστασία της ιδιωτικής ε, ζωής. Ως προς τις μυστικές υπηρεσίες, εμείς ε, θέλουμε να αλλάξουμε την νομοθεσία μας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες, περισσότερες επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κατασκοπίας. Έχουμε έρθει σε επαφή με εθνικές επιχειρήσεις επί του θέματος και χρειάζεται μεγαλύτερη, χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. το Υπουργείο Τεχνολογιών της Βραζιλίας έχει αναλάβει αυτό το ζήτημα. Όσο πιο πολύ ε, προχωρεί η τεχνολογία, τόσο περισσότερο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα χάσματα που δημιουργούνται. Ο πρόεδρος της ε, Γαλλίας, ο κύριος Ολάντ, ζήτησε ε, τη δημιουργία μιας συμφωνία την σύναψη μιας συμφωνίας εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ Βραζιλίας και Γαλλίας και εμείς προωθούμε τη νομοθεσία μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες και στο κράτος στα πλαίσια της συνεργασίας με το Μερκοσούρ. Θα πρέπει να προβάλλουμε αυτές τις αλλαγές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έμπρακτα αυτή τη συνεργασία. Ως προς τις ερωτήσεις σας, νομίζω ότι απάντησα. Θα ζητήσουμε να δημιουργηθεί και ένας οργανισμός, ο οργανισμός αντιμετώπισης της κατασκοπίας για την ε, προστασία του κυβερνοχώρου. Υπάρχει μια τέτοια διάρθρωση, αλλά είναι αρκετά ευάλωτη. Θα προτείνουμε τη σύσταση μιας προσωρινής επιτροπής, η οποία θα προτείνει μεταρρυθμίσεις ε, στη... και αναθεώρηση της νομοθεσίας μας, μέσα στα πλαίσια της ε, εξέτασης των δραστηριοτήτων κατασκοπίας. Ήδη ορισμένοι νόμοι, νομοθετήματα προωθούνται και άλλα βρίσκονται υπό μελέτη. Θα υποβάλουμε προτάσεις στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έτσι ώστε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προτεραιότητας κατά τον βραζιλιάνικο λαό. Μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης προστασίας που προβάλλουμε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα αυτοάμυνας και θα πρέπει να ε, δούμε πώς διαμορφώνεται και η νομοθεσία περί καλωδιώσεων, υπογείων καλωδιώσεων ή υποθαλάσσιων καλωδιώσεων που μας συνδέουν και με άλλες υπήρους. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Ο κύριος Φεράσο δεν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ο Ικάντος στο ξεκίνημα ανάφερε ρώτησε τις διαφορές σχετικά με την ε, Εξεταστική Επιτροπή για το ΕΣΕΛΟΝ. Εγώ θυμάμαι ότι και τότε ομοιότητα είναι ότι οι πληροφορίες που ζητούσαμε από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές δεν είχαν δοθεί. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η, δική η τωρινή έρευνα καλύπτει τα πάντα. Το ΕΣΕΛΟΝ ήταν πολύ μικρότερο Άλλη εποχή ήταν, το 2001 ήταν και πριν ε, την έκρηξη του ίντερνετ και τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στη ζωή μας, στη τεχνολογία. Αλλά ήταν εξαιρετική ε, η έρευνα τότε του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής ήταν ο Κάρλος Κοέλιο, Πορτογάλος και αυτός. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι για σας. Και άλλες ερωτήσεις τώρα. Η Κάρμεν Ρομέρο Λόπες και μετά ο κύριο Σαλαφράνκα και μετά ο κύριο Μπρόντς. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την πρόεδρο της ε, Βραζιλιάνική Εξεταστικής Επιτροπής της Γερουσίας. Ισπανίδα είμαι και θέλω να ρωτήσω για το ψήφισμα πλαίσιο που προτείνεται στον ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Το ψήφισμα αυτό τι θέλει να κάνει. Τι θέλετε εσείς να κάνετε με το ψήφισμα αυτό. Τι θέλετε να κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείες για το θέμα της παρακολούθησης αυτής. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε, και αυτό είναι μια πρόταση που σας κάνω, στην καταστροφή όλων των στοιχείων που λήφθηκαν παράνομα. Μπορεί να πετύχουμε κάτι τέτοιο που και τεχνολογικά είναι πολύ δύσκολο. Τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Μέχρι πού θα έφτανε η αστυνομική συνεργασία αν δεν υπάρχουν δικαστικές διαταγές που, ή αποφάσεις που αιτιολογούν την ύπαρξη των δεδομένων αυτών. Ο κύριος Σαραφράγκα και αυτός. Υπουργό τη Επιτροπή Εξωτερικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ καλησπέρα στην ε, γερουσιαστή Βανέσα, φίλη από πολλά χρόνια, από το Λατινοαμερικάνικο Κοινοβούλιο. Πολύ καλή ευκαιρία να, ξανα, να τα ξαναπούμε στα πλαίσια των ε, συνεδριάσεων της Επιτροπής αυτής, της Εκτασικής Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Έφτασα καθυστερημένα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Είχαμε επίσκεψη μελών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον είπα και τους ενημερώσαμε ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να κυρώνει ή να μην κυρώνει διεθνείς συμβάσεις που συνάπτει η Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για την κύρωση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και Επενδύσεων που συζητούμε αυτή τη στιγμή και που έχει μεγάλη σημασία για τα συμφέροντα και των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η γεωσιαστής μίλησε για τη σπουδαιότητα που έχει για τη Βραζιλία η υπογραφή των συμφωνιών ελευθερού εμπορίου. Εμείς εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να ακούσουμε κατά πόσον οι εταίροι σας στο Μερκοσούρ θα δεχθούν την βραζιλιάνικη πρόταση για τη διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΙΠΑ, σε τι βαθμό επηρεάστηκαν από την κατάσταση. Υπήρξε η, ανα... η... η... Ε, γεγονό ότι η πρόεδρος ε, των, της δεν επιτεψεύχε τελικά τη ΣΥΠΑ. έγιναν δεκτές, ε, έγινε δεκτή συγγνώμη από τη ΣΥΠΑ ε, ποιο ήταν το πλαίσιο που, μάλλον η, η μη επίσκεψη της Προέδρου το, της Βαζιλίας στη ΣΥΠΑ, τι επιπτώσεις είχε στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το γεγονός αυτό είχε αντίκτυπο όχι μόνο στο πλαίσιο των πολιτικών επαφών αλλά και στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και είπε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλόντς από την Επιτροπή Λίμπε. Πρόεδρε, στη Βρετανία οι επικεφαλείς των τριών υπηρεσιών ασφάλειας προσπάθησαν να περάσουν το μήνυμα ότι οι αποκαλύψεις βοήθησαν την ε, ε, τους τρομοκράτες και αύξησαν τον, τον, τον κίνδυνο ασφάλειας. Η επίσκεψη στην επιτροπή αυτή προσωπικό από την MI5 και το NSA μας διαβεβαίωσε ότι δεν κάνουν τίποτα που, που είναι βλαβερά για την ασφάλεια ούτε μπορούσαν να, οτιδήποτε μας αποκάλυπταν να έβλαπταν την ασφάλεια καταλήγετε κι εσείς το ίδιο συμπέρασμα για τις αποκαλύψεις τους, του κ. Σνόντεν. οι θέσεις αυτές των υπηρεσιών ασφάλειας κατά άποψή σας έχει στόχο να, να αμφισβητήσουν και να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του κυρίου Σνόντεν και άλλων ε, παρόμοιων ε, ατόμων μπορείτε να εξετάσετε στην ε, για ουσία της Βραζιλίας, ε, το ζήτημα αυτό να υπάρξει επίσημη απάντηση και να καταχωρηθεί ε, δημοσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Τους δίνω το λόγο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Constatações Εμείς στην δική μας εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή φτάσαμε σε ορισμένες διαπιστώσεις. Δεν έχουμε φτάσει στα, σε συμπεράσματα, αλλά θεωρούμε ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την NSA και όχι μόνο προσωπικών δεδομένων. Αυτό αποτελεί μία πρωταρχική ε, αλήθεια και καταδικάσαμε τη δράση των ΙΠΑ και ιδιαίτερα τη δράση της NSA. Άρα, στη Βόρειο Αμερική, από την Αμερική ε, υπάρχει μία αντίδραση διότι σε μια χώρα που προώθησε τη δημοκρατία, τον ιδιωτικό βίο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση και αυτό διαπιστώνουν οι κάτοικοι της ε, Βορειοαμερικής. Επίσης, ε, η τρομοκρατία ήταν μια σπίδα ήταν μία πρόφαση για να φτάσουμε σε πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα, επιχειρηματικού και ούτω καθεξής. Δηλαδή η δική μας η Petrobras αποτέλεσε αντικείμενο κατασκοπίας έτσι ώστε να ε, δοθούν πολλά στοιχεία για τους ε, διαγωνισμούς μας συμπεριλαμβάνοντας έναν μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος προκηρύχθηκε και επ' αυτού έγινε η καταγγελία ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλά στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο υποκλοπών. Δηλαδή η τρομοκρατία ε, χρησιμοποιείται ως πρόφαση για να ε, διαβρωθεί το σύστημα ασφάλειας και για να διαδοθούν πληροφορίες καθαρά οικονομικού χαρακτήρα ή να αποκαλυφθούν τέτοιες πληροφορίες. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυσκολίες με εσάς, διότι υπάρχει μία ε, υπεροψία, μία αλαζονία από πλευράς ΥΠΑ που θεωρούν ότι βρίσκονται πάνω από τον νόμο ότι μέσα στα πλαίσια της οικονομικής και στρατιωτικής διακυβέρνησης ε, κατέχουν ε, δεσπόζουσα θέση και έχουν μίζωνα λόγο, άρα βρίσκονται πάνω από όλα και από όλους. Δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζετε εσείς τα αντιμετωπίζουμε και εμείς. Το ψήφισμα υπαριθμών 4 των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα συμβολικό βήμα, καθαρά συμβολικό, από πλευράς κυβερνήσεών μας και από πλευράς της Ντίλμα Ρουσέφ, θεωρώντας ότι θα πρέπει να οριστεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο για να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε και να καταπολεμήσουμε την κατασκοπία και για να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε όρια, ούτε κριτήρια, ούτε αξίες που να υπερτερούν ως προς την ε, αμέριστη χρήση των ε, τεχνολογιών. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για χρήση ε, λογισμικού, αλλά για παραβίαση του ιδιωτικού βίου. Σε αυτά τα συμπεράσματα φτάνουμε στη χώρα μου. Επανεξετάζουμε το νομικό μας πλαίσιο θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία μας έτσι ώστε να ε, διευρύνουμε την προστασία. Η γερουσιαστής Βανέσα Γκρασιωτίν μίλησε για την χρήση του διαδικτύου, για την ομοθέσια που θα διέπει τη χρήση του διαδικτύου και μιλάμε γενικά για νέα στοιχεία, για το ότι ορίζουμε ε, ένα νέο πλαίσιο χρήσης του διαδικτύου. έτσι ώστε να έχουμε έναν ασφαλή ε, τρόπο επικοινωνίας σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, όπως το κατονομάζουμε. Θέλουμε λοιπόν να θεσμοθετήσουμε αυτές τις αξίες. Εμείς προσπαθούμε να ορίσουμε τώρα αυτό το πλαίσιο σε, αντίθετο, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήδη το 2001 αντιμετώπισε το σύστημα κατασκοπίας εσελών. Δηλαδή, εσείς από το 2001 μέχρι το 2013 είχατε μία ε, πιο προωθημένη εξελεκτική πορεία. Την Παρασκευή μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Γαλλικής ε, Δημοκρατίας, ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος εξέφρασε την αλληλεγγύη του με την πρόεδρό μας ε, Ντίλμα Ρουσέφ. Θέλουμε να δούμε πού ε, βρίσκονται τα ευάλωτα στοιχεία μας, πού είμαστε πιο ευάλωτοι και γι' αυτό ακριβώς παραβιάστηκε και το, ε, το πλαίσιο λειτουργίας και δράσης μας. Μας διέπουν φιλικές ε, σχέσεις. Ε, βεβαίως και η Ντίλμα Ρουσέφ είχε προσκληθεί από τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά αναβλήθηκε αυτή η επίσκεψη διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στα πλαίσια ενός ειλικρινούς διαλόγου. Αυτό ακριβώς είπαμε και στην πρέσβη των ΙΠΑ στη χώρα μας. Δηλαδή ότι η ΙΠΑ και ο Μπαράκ Ομπάμα θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις για να ξαναδούμε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Εμείς θεωρούμε ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι μας διέπουν σχέσεις φιλίας με τις ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε, και έχουμε και ένα ε, κοινό παρελθόν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η αντιμετώπιση της κατασκοπίας, να υπάρχει ασφάλεια στις επικοινωνίες αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μετά από αυτή τη γενικότερη διάγνωση, το διαγνωστικό ε, σκέλος, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Και ε, να επενδύσουμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κυβέρνο πόλεμο, κάτι που είναι μόνιμο και επίκαιρο. Ο κύβερνο πόλεμος, όπως και η παγκοσμιοποίηση, είναι κάτι διαφυσβήτητο και μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε και να κάνουμε μια σειρά, να υποβάλουμε μια σειρά συστάσεων προς την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για την αντικαταστροφοκοπία και στα πλαίσια της ανάγκης η χώρα μας να είναι αυτάρκης σε συστήματα προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις. Είναι βεβαίως ε, προφανές ότι πρέπει να δούμε την κατάσταση προσεκτικά γιατί η Γερμανία με εξαιρετικά σούπερ μοντέρνα συστήματα την ίδια ε, κατάσταση βίωσε. Το, ε, το τηλέφωνο της κυρίας Μέρκελ το παρακολουθούσαν από ό,τι ακούστηκε. Αν η Γερμανία δεν μπορεί να προστατευθεί από την παραβίαση αυτή πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Γι' αυτό πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας και υπολογίζουμε σε εσά το Κοινοβούλιο για να ε, υπάρξει ένα νέο πλαίσιο σεβασμού των ε, παραδόσεων και των, ε, του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεουσέστη, ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική και ουσιαστική συμπεριφορά. Ε, συνεισφορά. Ευχαριστώ λοιπόν ε, και τους δύο ε, σας, κυρία Γκρατσιωτίν, κύριε Φεράς. Δεν νομίζω πως έχει κάποιος ζητήσει το λόγο. Όχι, κυρία Γκόμες, έχετε κάποιο συμπληρωματικό σχόλιο. Ήθελα να ρωτήσω τους φίλους μας από την γερουσία της Βραζιλίας να μας μιλήσουν για τις εθημερείς συμφωνίες που έχει η Βραζιλία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Για παράδειγμα, τα PNR, Συμφωνία για τα Δεδομένα των Επιβατών ή κάποιες άλλες συμφωνίες ε, όπως εκείνες για την αντιτρομοκρατία. Σκέφτεστε τι επιπτώσεις έχουν οι ερευνές σας στις συμφωνίες αυτές. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ζητήσει αναστολή κάποιων συμφωνιών που είναι σε ισχύ, αναστολή, μέχρι να αποκτήσουμε ένα σαφές πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα δικά μας πρότυπα όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εσείς λοιπόν σκέφτεστε να αναλάβετε τέτοιες δράσεις όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, εξετάζουμε τις συμφωνίες αυτές, τις αναλύουμε. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα που να μας ε, οδηγήσει στο να ζητήσουμε αναστολή των εδημερών αυτών συμφωνιών. Χρειάζεται περισσότερη και εις βάθος ανάλυση προτού κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ε, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, αυτές δεν έχουν επηρεαστεί. Και η πρόεδρος το είπε αυτό ξεκάθαρα στο Κοινοβούλιο. Φυσικά και η εκτελεστική εξουσία έχει αναλάβει δράσεις, έχει συσταθεί διερευνητική επιτροπή, όμως ήταν σαφές ότι αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις ε, υπόλοιπες σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζεται να λάβουμε τα μέτρα που εμείς θεωρούμε σωστά, να φροντίσουμε ώστε να ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα και η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει λάβει μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Και έχουμε την υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη Διερευνητική μας Επιτροπή. Και το 2014, τον Απρίλιο, θα ξεχθεί ένα συνέδριο που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο γερουσιαστής Φεράσο μόλις ε, το είπε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικό στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό πλεονέκτημα και δύναμη και κυρίαρχη θέση ότι θα έχουν και το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις ε, διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Και Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι το 2001 το διαδίκτυο δεν είχε τις ίδιε δυνατότητε που έχει το 2013 τώρα και φανταστείτε πόσο πιο μπροστά θα μας φτάσει το 2023. Το διαδίκτυο πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και ε, της καθημερινής και της στρατιωτικής ε, ζωής και είναι αναγκαίο, απαραίτητο για όλου. Έτσι λοιπόν, καθώς ε, ορίζουμε το δικό μας πλαίσιο για αυτές τις ε, διμερείς συμφωνίες, πρέπει να φροντίζουμε ώστε να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα και οι πολίτες μας να έχουν την ίδια προστασία με τους ε, Αμερικανούς πολίτες. Και πιστεύουμε πως εμείς πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα στην δημιουργία τέτοιων συμφωνίων και με εσάς. Τώρα, όπως είπα, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και οτιδήποτε προέρχεται από εμάς και από εσάς θα είναι πιο ισχυρό εάν το πούμε με ένα στόμα. Θα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Πιστεύουμε λοιπόν πως πρέπει να τονιστεί η σημασία της συνεργασίας ημών και ημών. είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Και να σας πω ότι διερευνάται αυτή τη στιγμή το αίτημα ασύλου από τον Edward Snowden και πιστεύουμε πως μπορεί να του δοθεί Είναι μια μονομερής απόφαση από τη Βραζιλία. Δεν έχει καμία επίπτωση και δεν θα έπρεπε να έχει ε, στις σχέσει σχέσεις μας, εμπορικέ εμπορικές, τις ε, διπλωματικές, διότι η πολιτική της Βραζιλίας όσον αφορά το θέμα αυτό είναι να δίνεται άσυλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Εσεί στην Ευρώπη είστε πιο κοντά στη Ρωσία και αναρωτιέμαι ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση. Δεν ξέρω αν εσεί θα είχατε πιο εύκολο έργο του να, το να χορηγήσετε άσυλο στον Σνόουντεν. Μάλιστα, λέει πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνεισφορά σα και θα ήθελα να τελειώσω όπω αρχίσαμε, λέγοντα δηλαδή ότι υπάρχει εξαιρετική συμμετρία ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες πραγματικά. Και μάλιστα όταν αναφερθήκατε στο πρόγραμμα Echelon μου δώσατε την εντύπωση, με καθησυχάσατε, διότι ξέρω ότι ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάτε. Είστε απόλυτα ενημερωμένοι και πιστεύω πως ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να ξέρουν οι μη Αμερικανοί πολίτες πώς μπορούν να μηνθούν και πώς μπορούν να συμπεριφερθούν. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε αυτό το απόγευμα για αυτήν την βιντεοδιάσκεψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, uh, Ήταν... Είναι πολύ σημαντικό όμως να ακούσουμε και την απάντηση. Ε, από όσο γνωρίζω, λέει η κυρία Γκόμες, Ο κ. Νόμπεν δεν ζήτησε πολιτικό άσυλο επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν κάποια κινήματα, στη Γερμανία για παράδειγμα, θα μπορούσε να μας πει η κυρία Ζήπελ περισσότερα γι' αυτό, όπου οι πολίτες ζητούσαν από την κυβέρνησή τους να τους χορηγηθεί άσυλο. Δεν έχει ε, ζητήσει όμως επίσημα άσυλο ο Σνόντεν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα όταν συζητούσαμε το ενδεχόμενο να καλέσουμε τον Edward Snowden να καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω βιντεοδιάσκεψης, όταν αναφέραμε λοιπόν το ενδεχόμενο αυτό, οι Αμερικάνοι ε, απάντησαν ότι αυτό δεν θα το πάρουμε και τόσο θετικά. Ε, το αντίθετο μάλιστα, διότι ο, για μας ο Snowden είναι προδότης, δεν είναι κάποιος που έχει καταγγείλει παρατυπίες. Και φυσικά σημειώσαμε εμεί την αντίδρασή του αυτή. Η όμω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει αποφασίσει να τον ε, καλέσει ω μάρτυρα μέσω βιντεοδιάσκεψης. Σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Πραγματικά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό σα ευχαριστώ και το χρόνο σα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και του συναδέλφου ευρωβουλευτές που βρέθηκαν εδώ τόσο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση και του διερμηνεί. το χρόνο τους Κύριε Μπρόντσιν, έχετε να ρωτήσετε κάτι επί της διαδικασίας. Αν κατάλαβα καλά, η συνεδρίαση συνεχίζεται αύριο το πρωί. Η απόφαση όμως να διεξαχθεί η ακρόαση αύριο το πρωί ελήφθη χθε, όχι την περασμένη Παρασκευή, με συγχωρείτε. Και εγώ το έμαθα μόλις χθε. και άλλαξα. Δεν μπορούσα να αλλάξω τα εισιτηριά μου και ελπίζω να μην σας λείψω πάρα πολύ. Πάντως θα ήθελα να πω την επόμενη φορά να ενημερώνετε εγκαίρως για το πότε θα διεξαχθεί μια συνεδρίαση. Ναι, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο διαφανή γίνεται έτσι ώστε να έχουμε τη μέγιστη παρουσία εδώ, να έρχεστε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και είναι πολύ δύσκολο να διαβιβάζονται τα έγγραφα εγκαίρως. Υπάρχει και ένα άλλο έγγραφο που έχει καθυστερήσει από χθε, το οποίο μάλιστα είναι κάτι που είναι δική μου ευθύνη, την αναλαμβάνω. Αυτό έγινε απλά, μια καθυστέρηση. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε αύριο, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω όσον αφορά αυτό ότι η γραμματεία εργάζεται πραγματικά πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να δημιουργήσει το πρόγραμμα για αυτές τις ακροάσεις. Είναι πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο έχει χειριστεί το θέμα. Φυσικά όμως ε, αυτό συμπεριλαμβάνει και την όσο το δυνατόν και ρότερη ενημέρωσή σας. Θα το σημειώσουμε λοιπόν.